έρχονται αυτά στην συνολική μας πολιτική για να καταπολεμούμε τέτοια ε, ε, προβλήματα σε καιρούς οικονομικής ύφεσης και κρίσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ στον αδελφέ Τάνο, κλαίει ο Πρόεδρος. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την έκθεση Μάρτιν και τις επεξηγήσεις ψήφου. Όπως σας είπα προηγουμένως λοιπόν συνάδελφοι, θα διακόψουμε Μάλλον δεν θα μπορέσουμε να ακούσουμε τις επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση Μπουτικόφερ για την αναβιομηχάνηση γιατί θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα για την ε, σύνοδο που θα ξεκινήσει στις 3. Θα τις ακούσουμε λοιπόν αύριο, πέρας της ε, σύνοδου.